Τα πρακτικά και τα εγκριθέντα κείμενα της συνεδρίας 14, 14 Απριλίου είναι διαθέσιμα. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπάρχουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά της συνεδρίασης της 14ης Απριλίου. Γι' αυτό συζητάμε. Όχι, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Τα πρακτικά εγκρίνονται. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Όταν θα τελειώσουμε τις προκαταρκτικές διαδικασίες, τότε μπορείτε να πάρετε το λόγο. Κυρίες και κύριοι, Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων